Καλημέρα σας. Ε, μπορούμε σιγά σιγά να ξεκινάμε και για να σας φτιάξω λίγο τη διάθεση ε, δεν είδατε πως έφτασε ο κύριος Ντες. Ε, ήρθε με την καρτούλα του, την έβαλε μπροστά στη θέση του και μετά δεν είχε θέση να κάτσει ο άνθρωπος. Δεν ξέρω αν αυτό έχει κάποια συμβολική σημασία ή κάποιος έκανε δολιοφθορά, αφαίρεσε την <laughs> καρέκλα από τον κύριο Ντες. Εν πάση περιπτώσει. Ας ξεκινήσουμε. Οι διερμηνείς έχουν να μας διαβάσουν ένα μήνυμα, οπότε παρακαλώ φορέστε τα ακουστικά σας για να ακούσουμε το μήνυμα των διερμηνέων. Βρισκόμαστε στην ε, τρίτη εβδομάδα κινητοποιήσεων λόγω της εργασιακής διένεξης με τη διοίκηση για τις συνθήκες εργασίας μας. Σε ορισμένες καμπίνες έχουν επιστρατευτεί όλοι οι διερμηνείς και είναι υποχρεωμένοι να εργαστούν. Αυτό ουσιαστικά καταργεί το δικαίωμά του στην απεργία και συνιστά διάκριση προς τις υπόλοιπες γλώσσες. Ως εκ τούτου και σε ένδειξη αλληλεγγύης, η ελληνική καμπίνα δεν θα προχωρήσει στη στάση εργασίας που προβλεπόταν για τη σημερινή συνεδρίαση. Μάλιστα. Νομίζω ότι τα χειροκροτήματα μπορούν να κλειφθούν ως έκφραση υποστήριξης προς τους διερμηνείς. Σας ευχαριστούμε για την ανακοίνωση, λέει ο Πρόεδρος. Ε, φαίνεται αυτή η καθυστέρηση εκ μέρους της δίκησης δίνει την εντύπωση ότι έχει ξεκινήσει διακοπές θερινές.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 ιδιαίτερα και το λέω αυτό εμφατικά ιδιαίτερα για την πολύ καλή, την αγαστή συνεργασία που είχαμε με τους σκιώδεις εισηγητές. Ε, είχαμε, πετύχαμε πολλές καλές ε, συμβαστικές ε, προτάσεις και θέλω να σας μεταφέρω δύο μηνύματα. Το ένα είναι το ουσιώδης μήνυμα. Το μήνυμα είναι ότι η στόχοι που είχαμε το 2009 να επιτρέπεται η δυνατότητα κατάργησης γραφειοκρατίας ή ο στόχος της απλουστευσής, αυτός ο στόχος δεν έχει καν προσεγγιστεί, πόσο μάλλον επιτευχθεί. Γι' αυτό λοιπόν καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταθέσει ένα καινούριο κανονισμό μέσα σε 120 μέρες, να μπορεί ε, μία ε, δραστική ουσία να αδειοθωτηθεί. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι εύχομαι από τι πολλέ και καλέ σημαντικέ προτάσει που επιτύχαμε με τη συνεργασία των πολιτικών ομάδων. Εύχομαι ε, το πνεύμα αυτών των ε, συμβαστικών προτάσεων να υιοθετηθεί και από την Επιτροπή περιβάλλοντο. Και αυτό νομίζω ότι θα μπορεί να είναι ένα πολύ καλό δείγμα για τη συνεργασία ανάμεσα στι επιτροπέ. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όντως ε, πολύ φιλόδοξες αυτές οι ευχές, μακάρι να πραγματοποιηθούν. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά τη συμβαστική τροπολογία Α. Παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία για τη συμβαστική τροπολογία Α. Περιμένουμε μερικούς ε, συναδέλφους να ψηφίσουν την κυρία Εράνς Καρσία προκειμένου. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται η συμβαστική τροπολογία Α και περνάμε στη συμβαστική τροπολογία Β. Β. Β. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Πάμε στη συμβαστική Σ, λέει ο πρόεδρος. Συμβαστική τροπολογία Σ, τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία D, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας, λέει εγκρίνεται. Πάμε στην ε συμβαστική τροπολογία. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία F. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην τροπολογία 50. Ποιος είναι υπέρ, διανατάσσω στις χειρός, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 52. Ποιος είναι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Ο κύριος Άγνιου. Κύριε Πρόεδρε, ε, μου επιτρέπετε να σας διακόψω. Εδώ έχουμε κάποιον απόντα και το τηλέφωνο του συνέχεια χτυπάει και δημιουργεί φασαρία. Μπορεί κανείς παρακαλώ να το κλείσει, να το απενεργοποιήσει. Εγώ δεν έχω τέτοιες τεχνικές ικανότητες για να το διακόψω. Λυπάμαι που σας διακόπτω, αλλά νομίζω ότι εκνεύριζε τους πάντες αυτός ο θόρυβος. Κανά πρόβλημα. Τροπολογία 52 της κυρίας Μαγκίνης υπέρ επανάληψη. Ευχαριστώ. Εγκρίνεται. 54 Τις κυρίες Μαγκίνες και Ντελαέ. Εγκρίνεται. 55. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 56 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 57 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία G. G. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και πάμε στην τροπολογία 129. Διανατάσσεως της χειρός υπέρ. Εγκρίνεται. 103. Διακοπή. Η 129 εγκρίθηκε. 140 λέει πρόεδρος, υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 158 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία H, άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται και πάμε στην τροπολογία 14. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 16. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 17 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 18 υπέρ. Εγκρίνεται. 21 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 24 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 25 υπέρ. Κατά απορρίπτεται 26 υπέρ κατά απορρίπτεται 27 υπέρ κατά απορρίπτεται 28 υπέρ κατά απορρίπτεται 29 υπέρ κατά απορρίπτεται 30 υπέρ κατά απορρίπτεται συμβαστική τροπολογία I άρχιτη ψηφοφορία τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 66, διανατάσεις της χειρός, ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 68 υπέρ, κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος, άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 68. Τέλος. Απορρίπτεται. Καλώς που το ελέγξαμε. Τροπολογία 70. Ποιος είναι υπέρ. Κα... Κατά. Εγκρίνεται. 71. Υπέρ. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 70. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 71. Ποιος είναι υπέρ εγκρίνεται. 74 κατά τμήματα. Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα, ή μάλλον ηλεκτρονικός έλεγχος για το πρώτο τμήμα της 74. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 74 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 75. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 76 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία J. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 86 του κυρίου Νταντά. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 90. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία Κ. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. εγκρίνεται. Τροπολογία 92, Διανατάσσεω τη χειρός. Ποιο είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 94, Ποιο είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 90 96 Ποιος είναι υπέρ Κατά Απορρίπτεται 100 υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία L. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται και πάμε στην 109. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 112 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 114 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία μη. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία νη. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 125 του κυρίου Νταντά. Ποιος είναι υπέρ, εγκρίνεται. 127 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 128, ποιος είναι υπέρ, εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τη συμβαστική τροπολογία όμικρον υπέρ, ε, άρχιτη ψηφοφορία, συγγνώμη. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 143 τροπολογία, διανατάσσεως της χειρός υπέρ, εγκρίνεται. 145 υπέρ, εγκρίνεται. 147 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 149 υπέρ, εγκρίνεται. 152 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 154 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 155 υπέρ, εγκρίνεται. 157 υπέρ, εγκρίνεται. 159 υπέρ, εγκρίνεται. 161 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 162 υπέρ, κατά, ηλεκτρονικός έλεγχος για την 162. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας απορρίπτεται. 163 Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 164 υπέρ. Εγκρίνεται. 165 υπέρ. Εγκρίνεται. 167 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 168 υπέρ. Εγκρίνεται. 169 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Και ψηφίζουμε το σύνολο της γνωμοδότησης, όπως έχει τροποποιηθεί. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κύριε Σιγητά. Θέλετε το λόγο μήπως. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Όπως σας είπα, συμπεριέλευα πολλές καλέ ιδέες ε, τη επιτροπή μα στην γνωμοδότηση αυτή και τελειώνει εδώ αυτό. Εμεί ε, το τον συνάδελφο. Πάμε στο σημείο 4. Αξιοποίηση τη θάσευση τη παγκοσμιοποίηση, εμπορικέ πτυχέ. Αρμόδια καθήλια επιτροπή είναι η Επιτροπή Διεθνού Εμπορίου. Εμεί ε, συντάξαμε γνωμοδότηση, την οποία ανέλαβε η κυρία Κάντεμπαχ. Την ευχαριστούμε θερμά για την εκπόνηση της γνωμοδότησης. Ε, παρακαλώ, κυρία Κάντεμπαχ, για να μας κάνει μια εισαγωγή στην ψηφοφορία. Καλημέρα σας. Θέλω να ευχαριστήσω απλά τους συναδέλφους που έκαναν πολύτιμες ε, προτάσεις. Όλο αυτό το καιρό συζητούμε για τις προκλήσεις, τις ευκαιρίες αλλά και τους κινδύνους που ε, προέκυψαν από την παγκόσμια αγορά, ιδιαίτερα για τον ευαίσθητο τομέα της γεωργίας. Και ελπίζω πάρα πολύ η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή να λάβει υπόψη τα πάρα πολύ εύλογα ε, μελήματα και ανησυχίες των αγροτών και της υπαίθρου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Κάντεμπαχ. Οι εξωτερικοί παράγοντες επηρεάζουν όλο και περισσότερο τη γεωργία. Και σίγουρα εξωτερικές εμπορικές πτυχές ασκούν άμεση επίδραση στη γεωργία. Γι' αυτό και όλο και πιο συχνά συζητούμε αυτό το θέμα. Και καλό θα ήταν η, η Επιτροπή Εξωτερικού Εμπορίου να ασχοληθεί και με το θέμα αυτό. Γιατί χρειάζονται πολλά κονδύλια για το γεωργικό προπολογισμό και σίγουρα οι εξωτερικοί παράγοντες επηρεάζουν την κατάσταση τη γεωργίας. Ψηφίζουμε την τροπολογία 1, διανατάσσεω τη χειρό, είναι τη κυρία Κοτκέιτο. Ποιο είναι υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία A. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 11. Δυνατές τη χειρό υπέρ. Κατά. Σωστή παρατήρηση. Το επιβεβαιώνει και η γραμματεία. Λάθος το λέει ο κατάλογο. Πρώτα θα πρέπει να ψηφίσουμε την 8. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Πάμε τώρα στην τροπολογία 11, υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 12, υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 13, υπέρ, εγκρίνεται. 14, υπέρ, εγκρίνεται. 15, υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 16, υπέρ, εγκρίνεται. 17, υπέρ, εγκρίνεται. 18, υπέρ, εγκρίνεται 19 υπέρ εγκρίνεται 20 υπέρ κατά απορρίπτεται 21 ποιος είναι υπέρ εγκρίνεται 22 υπέρ εγκρίνεται συμβαστική τροπολογία β άρχεται η ψηφοφορία τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 34. Ποιος είναι υπέρ? Εγκρίνεται. 39 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία C. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 41. Διανατάσσεως της χειρός. Ποιος είναι υπέρ, είναι η τροπολογία Αγγιλέρα. Κατά. Απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 41. Άρχεται η ψηφοφορία. Πρόκειται για τροπολογία της κυρίας Αγγιλέρα, όπως είπαμε. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Λυπούμε, λυπούμε, έκανα λάθος, λέει ο πρόεδρος. Ζητώ, συγγνώμη. Όταν ψηφίζουμε ε, με τα χέρια και είδα τους συντονιστές, ε, δεν κατάλαβα το αποτέλεσμα. 42, ποιος είναι υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. 43. Ηλεκτρονικός έλεγχος και για τη 42, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται αυτή. Ε, πραγματικά, αν και αυτή τη φορά έκανα λάθος, θα ήμουν απαρηγόρητος. 43. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 44. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 44. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 45 υπέρ. Εγκρίνεται. 46 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 46. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία D. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία ε. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. εγκρίνεται. Τροπολογία 58 του κυρίου Καπούτο. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 59 υπέρ. Εγκρίνεται. 61 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 63 υπέρ. Εγκρίνεται. Αλλά στο λέξουμε. καλό κακού. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 63, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 64, υπέρ. Εγκρίνεται. 66. Ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 67 υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος για την 67 έρχεται η ψηφοφορία τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται τροπολογία 68 ποιος είναι υπέρ κατά απορρίπτεται Συμβαστική τροπολογία F, άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται και πάμε στην συμβαστική τροπολογία G, άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 82. Ποιος είναι υπέρ? εγκρίνεται. 84 υπέρ κατά απορρίπτεται. 86 υπέρ κατά εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία H. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. εγκρίνεται. Τροπολογία 96. Νταντάν και Ντελαϊέ. Ποιος είναι υπέρ? Εγκρίνεται. Τροπολογία 97. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία I. Λιώτα, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 104 των Ισπανών φίλων μας. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 105. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία J. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πάμε στη συμβαστική τροπολογία K. Άρχεται η ψηφοφορία. Zamykam głosowanie. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 109. Διανατάσσω τη χειρός. Απορρίπτεται. 113 υπέρ. Εγκρίνεται. 114 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 114. Άρχεται η ψηφοφορία. 114. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 115 δεκαπέντε. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική λάμδα. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. εγκρίνεται. Τροπολογία 120. Ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία μη, Άρχιτε ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία νη. Άρχιτε ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. 122 ψηφίζουμε ποιος είναι υπέρ, κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος, άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 122. Τέλος ψηφοφορίας. εγκρίνεται. 123. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 124. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 125 υπέρ εγκρίνεται. 126 υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία τέλος ψηφοφορίας απορρίπτεται και το σύνολο της γνωμοδότησης ε, μαζί με τις τροπολογίες άρχεται η ψηφοφορία παρακαλώ Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεν ξέρω αν η συγγήτρια την οποία συγχαίρομαι καθώς και του συνεργάτες της. Δεν ξέρω αν θέλει το λόγο, κυρία Κάντεμπαχ. Θέλετε το λόγο. Τον έχετε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους. Τώρα το θέμα είναι και οι συνάδελφοι της Επιτροπής Ίντα, ε, τα δικά μας μέλη δηλαδή που είναι και στην Ίντα, να διαφημίσουν την έκθεση και να φροντίσουν την ομοδότηση καλύτερα, να φροντίσουν να συμπεριληφθούν όλα αυτά στην έκθεση της Ίντα. Σας συγχαίρουμε και ενστερνιζόμαστε την ευχή σας. τον Σεπτέμβριο θα ψηφίσει η αρμόδια καθήλη επιτροπή, τον Οκτώβριο θα πάει στην Ολομέλεια. Ε, να καλωσορίσω και τους ε, καλεσμένους. Ε, βέβαια παρακολουθείτε τις εργασίες μας σε μια τεχνική φάση ε, της συνεδρίασης, την φάση της ψηφοφορίας ενώ το απόγευμα θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Επίτροπο Ανδριου Κάιτες. Πάντως σας καλωσορίζουμε στη συνεδρίαση. Περνάμε τώρα στο σημείο 5. Η συγητή της γνωμοδότησης είναι ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. Βαλκάρσελ Σίσο. Αρμόδια κατ' ουσίαν είναι η Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εμείς ε, εκπονούμε γνωμοδότηση για την εντολή ε, για τον τριμερή διάλογο για τη δημοσιονομική διαδικασία. Αποουσιάζει ο κύριος Αντιπρόεδρος, αλλά μπορώ να σας πω και εγώ δύο λόγια. Όπως σας είπα, πρόκειται για γνωμοδότηση που θα χορηγήσουμε στην Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια κατ' ουσία. Η συγγετής μας είναι ο κύριος Βαλκάρσελ Σίσο. Ε, κατατέθηκαν 44 τροπολογίες, συντάχθηκαν και συμβαστικές τροπολογίες 4, 5, από τον εισηγητή και νομίζω δεν έχω να πω τίποτα άλλο σε αυτή τη φάση. Δεν ξέρω αν κάποιος θέλει το λόγο. Α, κυρία Μόγα. Αντικαθιστά τον κύριο Ντενανό. Συγγνώμη που έκανα λάθος την προφορά αρχικά. Θέλω να μάθω πρώτα το όνομά σας ευελπιστούμε ότι θα έχουμε πολύ αγαστή συνεργασία μαζί σας, όπως είχαμε και με τον κύριο Ντενανό. Και δεν ξέρω αν θέλετε το λόγο, πολύ ευχαρίστω. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όντω είναι βαρύ το καθήκον που μου αναλογεί να αντικαταστήσω τον κύριο Ντενανό που είχε την καλοσύνη να μου παραχωρήσει ένα χρόνο τη θητεία να σας αναφέρω τι έγινε στη συνεδρίαση. Ήταν πάρα πολύ θετικό το κλίμα. Η γνωμοδότηση συζητήθηκε χωρίς να υπάρξει μεγάλη αντίρρηση. Το έγγραφο τώρα είναι στα χέρια της Επιτροπής Προϋπολογισμού ε, για να ψηφίσουν τον προβλέψιμο του 2019 και θα ξαναγυρίσει σε μας. Όλα καλά λοιπόν, μεγάλη νυφαλιότητα επικρατεί. Σας ευχαριστούμε. Όντω, είναι πολύ ενδιαφέρον το κοινοβουλευτικό έργο, γιατί ιδιαίτερα στην τελική ευθεία υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση εργασιών. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στην θητεία σας και είμαι σίγουρος ότι θα συνεργαστούμε. Περνάμε τώρα στην ψηφοφορία της γνωμοδότησης του κυρίου Βαλκάρσελ. Συμβαστική τροπολογία 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλο ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Τον Λουαζό και Κολομπιέ. Ποιος είναι υπέρ. Υπέρ. Κατά απορρίπτεται. Τροπολογία 7 του κυρίου Καπούτο υπέρ εγκρίνεται. Τροπολογία 10 υπέρ κατά απορρίπτεται. Τροπολογία 8 της κυρίας Μαγκίνες. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 11. Υπέρ εγκρίνεται. 13 του κύριου Βιέγκας υπέρ εγκρίνεται. 14 υπέρ εγκρίνεται. 15 υπέρ κύριο με και Φέντερλε. Υπέρ 15 κατά. Απορρίπτεται 16 υπέρ. Εγκρίνεται 17 υπέρ. Εγκρίνεται 18 υπέρ. Εγκρίνεται 19 υπέρ. Εγκρίνεται. 20 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 21 υπέρ. Εγκρίνεται. 22 υπέρ. Εγκρίνεται. 23 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 24 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 25 υπέρ. Κατά απορρίπτεται 26 υπέρ κατά απορρίπτεται 27 υπέρ κατά απορρίπτεται 29 υπέρ εγκρίνεται 29 το κύριο Μπούτα ε, εγκρίνεται είπαμε Συμβαστική τροπολογία 2 άρχεται ψηφοφορία Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται συμβαστική τροπολογία 3. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται τροπολογία 33 του κυρίου Βιέγκας. Ψηφίζουμε δυνατές χειρός υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 34, Χόισλινγκ υπέρ, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 4, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 42. Ποιος είναι υπέρ? Εγκρίνεται. Και 43 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. και ψηφίζουμε το σύνολο της γνωμοδότησης όπως έχει τροποποιηθεί. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται και συγχαίρομαι τον κύριο Βαλκάρ Σελσίσο. Παρακαλώ διαβιβάστε το τα συγχαρητήριά μας. Ολοκληρώσαμε τις ψηφοφορίες. Περνάμε τώρα στο σημείο 6 της ημερήσιας διάταξης, Παρασκευή και θέση εμπορία φαρμακούχων ζωοτροφών. Κατάργηση της ε, οδηγίας του Συμβουλίου 9 167. Η συγκεκριά μας είναι η κυρία Αγγιλέρα. Εμείς είμαστε αρμόδια κατ' ουσίαν επιτροπή ενώ γνωμοδοτήσεις ε, θα συντάξουν οι επιτροπές περιβάλλοντος, ο φίλος ε, Νόρμπερτ Λίνς. Ε, η ΙΜΚΟ αποφάσισε να μην συντάξει γνωμοδότηση και γνωμοδότηση επίσης θα συντάξει και η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων ενώ όπως είπα η συγκίτρια της έκθεσής μας είναι η κυρία Αγγιλέρα Α, γιατί αποσιάζει, λέει πρόεδρος, αλλά δεν την είδε. Α, συγγνώμη, χίλια συγγνώμη, δεν σας είδα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλους σας. Καλημέρα, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Πολύ επίκαιρο αυτό το θέμα σήμερα στην ημερήσια διάταξη. Εχθές έγινε ο τριμερής διάλογος που κατέληξε σε συμφωνία. Επιτέλους, σε αυτή την ε, συμφωνία για τον κανονισμό για τις φαρμακούχες ζωοτροφές. Εμείς τα διεκπαιρεώσαμε πάρα πολύ γρήγορα, αλλά μετά θυμάστε τι έγινε. Είναι ένας κανονισμός που είμαστε εμεί αρμόδιοι επί τη ουσίας, αλλά συνδέεται πάρα πολύ με τον κανονισμό για τα κτηνιατρικά φάρμακα, που είναι αρμόδια επί τη ουσίας η Επιτροπή Περιβάλλοντος. Και εκείνη τελείωσε τον τριμερή διάλογο. Και η Επιτροπή Γεωργίας και η Επιτροπή Περιβάλλοντος. Ο στόχος ε, που επετεύθη ήταν ε, ο επιθυμητός για όλους, δηλαδή εναρμόνιση στη χρήση, ε, παρασκευή και διανομή και κυκλοφορία στην αγορά των φαρμακούχων ζωοτροφών, είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταπολεμηθεί η αντοχή στα αντιβιωτικά. Στέλνουμε πολύ σημαντικά μηνύματα και συστάσεις από το Κοινοβούλιο και πετύχαμε αυτό που θέλαμε. Όλες οι χρήσεις, όλες οι χρήσεις για τις ζωοτροφές για τη διατροφή των ζώων και για τα φάρμακα που χορηγούνται για τη θεραπεία τους ρυθμίζονται με νέους κανονισμούς και στη συνέχεια καταξοδότηση πράξη για την χορήγηση από το στόμα των φαρμάκων. Και μέχρι τέλους εργαστήκαμε έτσι ώστε να συμπεριληφθούν κάποια στοιχεία στον κανονισμό. Δηλαδή, όταν πρόκειται για τρίτες χώρες που έχουν συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να υπάρχει ένα πολύ σημαντικό άρθρο αυτό το λέει στο 122 του κανονισμού για τα κτηνιατρικά φάρμακα, ότι υπάρχουν προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πρέπει να τηρούνται και από τις τρίτες χώρες για τη διατροφή των ζώων και τη χορήγηση φαρμάκων σε αυτά. Είναι μεγάλη ικανοποίησή μας ε, για την επιτυχία αυτή και επιτέλους, ε, ξανά και τελειώνω με τη συμφωνία αυτή, έχει μεγάλη σημασία Απαγορεύεται η προφυλακτική ε, χορήγηση αντιβιωτικών ή προληπτική χωρίς να στενούν τα ζώα. Ε, στόχος του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής μας ήταν να συμπεριληφθεί αυτό στον κανονισμό ε, για τα κτηνιατρικά φάρμακα και τις φαρμακούχες ε, ζωοτροφές. Είναι δύο κανονισμοί, επαναλαμβάνω, παράλληλη η διαπραγμάτευση και οι δύο συμφωνίες θα πρέπει να φτάσουν στην επόμενη Ολομέλη. Καλά, επόμενη τον Οκτώβριο νομίζω προβλέπεται να ψηφιστεί στην Ολομέλεια. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις εισηγητές, τους τεχνικούς, τη γραμματεία. Άντε μας Μανσέγο που έφυγε και μας ε, βοηθούσε μέχρι τέλους. Να ευχαριστήσω και τη Μάγκη, τη ε, βοηθό της σοσιαλιστικής ομάδας και τη Μαγδαλένα, την προσωπική μου βοηθό. Ήταν πάρα πολύ τεχνικός ο, οργανισμό, ο κανονισμός συγγνώμη, και αν δεν είχαμε όλη αυτή τη στήριξη δεν θα μπορούσαμε να τα ε, καταφέρουμε. Όλες οι πολιτικές ομάδες. Και αυτός ο στόχος δεν είναι της δικής μου πολιτικής ομάδας, είναι γενικός στόχος να καταφέρουμε αυτή η καταπολέμηση των αντιβιωτικών να περάσει. Να σταματήσει η χρήση από τη διατροφή και η χορήγηση από το στόμα φαρμάκων ουσιαστικά με την τροφή προληπτικά. Ευχαριστώ λοιπόν όλους τους τεχνικούς, όλους τους εμπειρογνώμονες και όλους τους ηγητές. Ευχαριστώ πολύ. Czy mamy jakieś zgłoszenia? Mr. Buda. Ποιος θέλει το λόγο από τους συναδέλφους, ο κύριος Μπούντα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να είμαι πολύ σύντομος. Θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Γκιλέρα για την προσπάθεια που κατέλαβε, κατέβαλε. Είναι μια τεχνική φύσεως έκθεση, πάρα πολύ δύσκολη. Νομίζω όμως ότι καταλήξαμε σε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Και θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι ε, η έκθεση αυτή και τα αποτελέσματα αυτά πρέπει να εφαρμόζονται σωστά. Γιατί στην Ολλανδία, παραδείγματο χάρη, υπήρχαν παραβιάσει του δικαίου. Χρησιμοποίησαν απαγορευμένε ουσίε, παραδείγματο χάρη, κατά την παραγωγή αυγών. Υπάρχουν λοιπόν πολλά, ειδήσει νέα σχετικά με αυτό. Προσπαθούμε να καταβάλουμε προσπάθειες, αλλά δεν καταλήγουμε πάντα σε καλό αποτέλεσμα, γιατί σα λέω δεν υπάρχει σωστή εφαρμογή αυτής ε, αυτών των απόψεων. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Ε, άλλος κάνει το λόγο. Όχι, από ό,τι βλέπω. Οπότε έχουμε την ευκαιρία να ξαναδώσουμε το λόγο στην κυρία Γιλέρα. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο. <laughs> Αυτό που έχει σημασία είναι να εναρμονιστούν οι δύο ε, αυτοί οι κανονισμοί και η γενική νομοθεσία να προσαρμοστεί. Ήταν πάρα πολύ απαραίτητο αυτό για να δώσουμε το καλό παράδειγμα ε, οι εκμεταλλεύσεις ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ε, Σας ευχαριστούμε. Μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο τότε. Το σημείο 7 που αφορά την παρουσίαση της έκθεσης της αποστολή της Επιτροπή Γεωργίας στη Φιλανδία. Να πω εισαγωγικά δύο λόγια. Ε, μια αποστολή της, της Επιτροπής μας ε, μετέβη 7 με 9 Μαΐου 2018 στο Κάινο στη... και τη Βόρεια Σαβωνία της Βόρειο-Ανατολικής Φιλανδίας χάρη στην αποστολή αυτή είχαμε την ευκαιρία να ε, δούμε από κοντά τις ιδιαιτερότητες ε, της φιλανδικής γεωργίας. Επισκεφθήκαμε πολλές διαφορετικές ε, γεωργικές εκμεταλλεύσεις και φάρμες και είδαμε πόσο περίπλοκη είναι η άσκηση γεωργικής δραστηριότητας σε περιοχές με πολλούς φυσικούς περιορισμούς και πόσο πολύπλευρη είναι. Ευχαριστούμε θερμά για τη διοργάνωση. Επίση ε, η αντιπροσωπεία μας επικεντρώθηκε στα θέματα βιοοικονομίας και ε, δάσοκομίας, γιατί πάνω από 70% της, ε, εκ, φιλανδικής καλύπτεται από δάση και είναι σημαντική πηγή και οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας τα δάση στη Φιλανδία. Υπάρχει πολύ στενή αλληλεπίδραση γεωργίας και δασοκομεία στην Φιλανδία. Επίσης ε, είδαμε ε, πολύ ενεργό και βιώσιμη διαχείριση των δασών στην πράξη. Είδαμε μια μεγάλη βιοπικιλότητα των δασών στη Φιλανδία και επίσης επισκεφθήκαμε ε, ιδιαίτερα καινοτόμες ε, εγκαταστάσεις ε, παραγωγής βιομηχανικών, ε, βιολογικών προϊόντων. Ε, πήγαμε και σε μια εγκατάσταση παρασκευής βιοκαυσίμων. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα από κάθε άποψη αυτή η αποστολή. Και γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την κυρία Έλση Κατάιναν για την άρτια διοργάνωση αυτής της αντιπροσωπείας. Καταφέραμε να επικεντρωθούμε σε πολύ ουσιαστικά θέματα. Ήταν πολύ μεστή, ε, μεστό το πρόγραμμα της αποστολής. Και αυτό, γι' αυτό ευχαριστούμε και πάλι θερμότατα την κυρία Κατάιναν για την οργάνωση. Έχει το λόγο πρώτα η κυρία Κατάινεν και μετά αν θέλουν και τα μέλη της αποστολής. Thank you, Mr. Ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε για τα πολύ ζεστά σας ε, λόγια και θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τη γραμματεία της Επιτροπής αλλά και όλους τους ε, συναδέλφους που συμμετείχαν σε αυτήν την ε, αντιπροσωπεία που μετέβη στη Φινλανδία. Η αντιπροσωπεία επισκέφθηκε τις περιοχές μας, το Υπουργείο μας, ε, τους γεωργούς επιτόπου και όλοι αυτοί περίμεναν την αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου. Εξάλλου αυτή η επίσκεψη ε, προβλήθηκε ιδιαίτερα στα μέσα ενημέρωσης της ε, Φινλανδίας. Πήγαμε και στη δική μου την περιοχή η οποία ασχολείται κυρίως με το γαλακτοκομικό και το Κάινεν το οποίο είναι πολύ γνωστό ε, για τα δάση του γενικότερα για τη φύση που υπάρχει εκεί. Τα ταξίδια διήρκεσαν πάρα πολύ γιατί η χώρα μας είναι είναι αραιοκατοικημένοι, αλλά είδαμε τουλάχιστον πολλά δάση και ε, λίμνες και όπως μας είπε και ο πρόεδρος, ε, πάνω από το 70% της χώρας μας ε, καλύπτεται από δάση και έχουμε και χιλιάδες λιμνών ε, σε πάρα πολλές περιοχές είδαμε ότι στην πλέον γεωργική χώρα του, του κόσμου, ο, η άνοιξη είναι περίπου λιγάκι σαν το χειμώνα. Το πρώτο θέμα και ίσως και το πιο εξωτικό ε, που αφορά στο πρόγραμμα ήταν η επίσκεψη στην ε, γεωργική εκμετάλλευση Ρέντια. Εκεί η συζήτηση περιστράφηκε συγκεκριμένα γύρω από τρία θέματα ε, για, τα, ε, για τους ε, λύκους και βεβαίως τα ελάφια, η τάρανδη. Αυτή είναι ιδιαίτερα έντονη η παρουσία τους στη Φινλανδία. Σε αυτό το ταξίδι, μεταξύ άλλων, συναντηθήκαμε συναντηθήκαμε και με τον πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης ε, Γεωργικών, Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων, τον κύριο Χαμάρτιλαν, τον Υπουργό Γεωργίας και Δασών. Επίσης, ε, επισκεφθήκαμε και ένα εργοστάσιο επεξεργασίας του ξύλου ε, όπου ε, γίνεται και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Προφανώς και πρόκειται για ανανεώσιμη πηγή ενέργειας και ο στόχος ε, της επισκέψης είναι να δούμε πώς τα πριονίδια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή βιοεθανόλης και ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης, επισκεφτήκαμε το Πόνσε, είναι ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές ε, μηχανημάτων στον κόσμο. Είδαμε επίσης ε, συγκεκριμένα πώς γίνεται η διαχείριση των δασών στη Φινλανδία και με τη χρήση σύγχρονων τεχνικών. Το 70% της ε, γης καλύπτεται από δάση. ω ως εκ τούτου θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η βιοπικιλότητα και η διάρκεια επιβίωσης, αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, είναι καθήκον όλων μας σε σχέση με τα δάση. Επισκεφτήκαμε και τα κεντρικά γραφεία και τις εγκαταστάσεις παραγωγής της Πόνσεν. Επισκεφθήκαμε το εργοστάσιο, εκεί είχαμε πολύ συγκεκριμένες εξηγήσεις που μας ε, ε, δόθησαν για το πώς ακριβώς κατασκευάζονται οι ε, μηχανές συγκομιδής. Επισκεφτήκαμε και μια γαλακτοπαραγωγική μονάδα ε, από τη διαχειρίζεται ένα ζευγάρι ε, με πάρα πολλές ε, υπομονάδες, 68 περίπου 68 γελάδες περισσότερο και όχι μονάδες παραγωγής. Την τελευταία μέρα είχαμε τη δυνατότητα να επισκεφτούμε μπορούσαμε να επισκεφτούμε μία από τις μονάδες στην ε, Φινλανδία όπου υπάρχουν, ε, ε, χρησιμοποιούνται συστήματα αυτοματισμού και ρομπότ. Και το τελευταίο κομμάτι του ταξιδιού μας αφορούσε τον αγροτουρισμό. Είναι μία οικογενειακή μονάδα Επισκεφθήκαμε και τις λίμνες το να κολυμπήσει κανείς ε, σε μία λίμνη το βράδυ. Ε, Βεβαίω ε, ήταν και αυτό μέσα στο πρόγραμμα. Αυτά εν ολίγης, πολύ σύντομα, μία περιγραφή της, του ταξιδιού μας που ελπίζω να βοήθησε στο να γίνει κατανοητό πως υπάρχουν διαφορετικές μορφές γεωργικών εκμεταλλεύσεων και ζωοτεχνίας στις διάφορες περιοχές της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε και πάλι θερμά για την οργάνωση αυτής της αποστολής. Ο κύριος Ντόρφμαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επί της δεν έχω να προσθέσω τίποτα. Συμφωνώ με αυτά που είπατε και εσείς Πρόεδρε. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον το ταξίδι αυτό. Ιδιαίτερα το σκέλος της δασοκομείας με ενδιαφέρει πάρα πολύ και ιδιαίτερα οι καινοτομίες ε, στο τομέα της δασοκομείας. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ τη συνάδελφο Κατάινεν για την εξαιρετική προετοιμασία ε, και όλη την πλαισίωση κατά τη διάρκεια του ταξίδιου. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε, κύριος Γιάρ. Yes, thank you, Chair, and I would like to... Uh, Κύριε Σχόιτεμα, ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την ΕΣΚ και την ε, ομάδα της για τη διοργάνωση αυτού του ταξιδιού στην αρχή πραγματικά με κατέπληξε η φιλοξενία των φυλαδών και η ομορφιά της χώρας. Ορισμένοι λένε που είναι το δάσος, παντού είναι δάσος, ολούθε. Και για μας είναι πολύ εντυπωσιακό για τη χώρα μου τις κάτω χώρες που έχουμε πολύ μικρές επιφανείς με δάσο. Και επίσης βλέπω πώς ε, ε, γίνεται η διαχείριση των δασών ε, αναδασώνονται ε, τα δάση που υλοτομούνται. Ορισμένοι λένε ότι κόβεται τα δέντρα για παραγωγή βιοκαυσίμων και μειώνεται το δάσος καθόλου. Αυξάνεται το δάσος ε, με την αναδάσωση. Και είναι καλή η παραγωγή ξυλίας, αλλά και πάρα πολύ βιώσιμη παραγωγή ενέργειας. Πολύ ενδιαφέρον για μένα. Και κάτι άλλο που με εξέπληξε, είναι το μεγάλο, τα μεγάλα σύνορα με τη Ρωσία πολύ μικρή ε, ε, περίοδος καλλιέργειας και παραγωγής. και είναι πολύ δύσκολο για τους αγρότες να παραμείνουν ανταγωνιστικοί ε, στην ευρωπαϊκή αγορά. Όσοι έχουν επιχειρηματικό πνεύμα και δυνατότητα υιοθέτηση νέων τεχνολογιών για να παραμείνουν λίγο πιο ανταγωνιστικοί. Αυτό μας δείχνει όμως ότι θα πρέπει να κάνουμε συζήτηση εδώ για την κοινή γεωργική πολιτική για τις πιο αεροκατοικημένες περιοχές ε, και ε, για τις περιοχές που έχουν πολύ μικρή καλλιεργητική περίοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Didn't go on that. Ο κύριο Άγνιο. Εγώ δεν πήγα σε αυτή την ε, αποστολή. Θα ήθελα όμω να πάω γιατί ήταν πάρα πολύ καλά οργανωμένη από ό,τι άκουσα. Το 2009 ε, σε όλη τη Φινλανδία από πάνω μέχρι κάτω στην ανατολική πλευρά και πρέπει να σας πω ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον το οδικό δίκτυο ε, υπάρχει ένα πολύ καλό οδικό δίκτυο αλλά στα σύνορα προς τη Ρωσία δεν υπήρχε σχεδόν κανένας οδικός χάρτης και γι' αυτό και εγώ και η γυναίκα μου δεν μπορέσαμε να το καταλάβουμε αυτό η Φινλανδία είναι μια χώρα ε, που μπορεί κανείς να ζήσει πάρα πολύ καλά από αυτή την πλευρά, γιατί από την άλλη πλευρά προς τη Ρωσία τα πράγματα είναι τραγικά. Ε, θα ήθελα να ρωτήσω, η επεξεργασία σαχαρότευλων εξακολουθεί να υπάρχει στη Φιλανδία, γιατί υπήρχε, αλλά δεν ξέρω τι ακριβώς ε, γίνεται σήμερα. Κύριε Κατάιν, θέλετε να απαντήσετε στην απόρία του κυρίου Άγνιου. Μπορείτε αμέσω να το κάνετε. Κοιτάξτε, θα απαντήσω στα φινλανδικά και θέλω να πω το εξή Στη Φινλανδία Όσον αφορά την επεξεργασία των σακαρότευτλων, ε, λίγες μονάδες έχουν απομείνει, διότι έχει υποβαθμιστεί αυτή η βιομηχανική μονάδα. Ε, σε λίγες μόνο περιοχές υπάρχουν κάποιες μονάδες ε, μεταποίησης και επεξεργασίας των σακαρότευτλων. Μία τελικά, όχι λίγες, μία. Μία είναι. Τα τελευταία λοιπόν χρόνια πραγματικά υπάρχει μία υποβάθμιση αυτού του κλάδου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους αδέλφους που συμμετείχαν σε αυτό το ταξίδι, σε αυτήν την προσωπία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια και ελπίζουμε να επανέλθετε σύντομα στο μέλλον στη Φινλανδία. Δεν βλέπω να θέλει άλλος κανείς το λόγο. Οπότε να πω ότι όλες οι εμπειρίες που αποκομίσαμε στη Φιλανδία θα τις εντάξουμε στη, στο καθημερινό μας έργο. Κοίτα, πολύ σημαντικό και αυτό το, το στοιχείο που αφορούσε τις ρωσοφιλανδικές σχέσεις. Και τι κάνει η Φιλανδία για τις βαλτικές χώρες γιατί έχει πολλές διασυνδέσεις ε, με τις βαλτικές χώρες. σίγουρα η καλλιεργητική περίοδος ε, διαρκεί πολύ λίγο, αλλά έχει πολύ πλούσιους ε, υδάτινους ορίζοντες. Η Φιλανδία υπάρχει πολύ νερό και είναι σημαντικό. Βοηθάει αυτό και την παραγωγή, κυρίως τη γάλακτοπαραγωγή. Αυτή, αυτά τα μεγάλα αποθέματα, είδα τόσο που έχει η Φιλανδία. Ε, είχαμε στην Επιτροπή μας ε, και Έλληνα συνάδελφο και τον εθάρρυνα να συμβάλλει στην σύσφυξη των σχέσεων Φιλανδίας-Ελλάδας Ε, συνεχάρημε λοιπόν την κυρία Κατάινεν, αλλά να συγχαρούμε και τους συνεργάτες της. Βλέπω εδώ κάποιος στην αίθουσα, γιατί πραγματικά ήταν το επιτελείο της κυρίας Κατάινεν ε, πολύ δραστήριο, πολύ αξιόλογη προσπάθεια που έκανε και διοργάνωση και ευχαριστούμε θερμά τους συνεργάτες της κυρίας Κατάινεν. Και μέσω ημών μπορούμε να ευχαριστούμε και την υπόλοιπη ομάδα. Ευχαριστούμε την κυρία Κατάινεν, ολοκληρώνουμε αυτό το σημείο. ολοκληρώνουμε τη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Γεωργίας αυτή τη στιγμή. Πολύ γρήγορα διεκπαιρεώσαμε το πρωινό τμήμα γιατί ψηφίσαμε σχετικά γρήγορα. Διακόπτουμε τώρα και στις μισή θα ξεκινήσουμε τη συνεδρία των συντονιστών, λίγο νωρίτερα από ό,τι προβλεπόταν, γιατί έχουμε έναν ε, μακροσκελή κατάλογο σημείων στην ημερήσια διάταξη. Οπότε καλό θα ήταν να ξεκινήσουμε νωρίτερα γιατί θα έχουμε πολλές συζητήσεις. Δεν μπορούσαμε να επισπεύσουμε ακόμη περισσότερο, μάλλον 11 παρατέταρτο θα ξεκινήσουμε τελικά. 11 παρατέταρτο γιατί δεν μπορούν νωρίτερα όλοι οι συντονιστές. Και μην ξεχνάτε ότι το απόγευμα θα ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση στις 2.30 με πρώτο σημείο την ανταλλαγή απόψεων με τον Επίτροπο. Οπότε παρακαλώ να είστε παρόντες για να μην μιλά ο Επίτροπος σε άδεια αίθουσα. Διακόπτουμε λοιπόν τώρα μέχρι τις 11 παρατέταρτο που θα ξεκινήσει η συνεδρίαση των συντονιστών και για τους υπόλοιπους ραντεβού στις 2.30 για την δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής.